Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφων. Έξι. Έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κ. Νικόλας Κόντης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κ. Κουντής, συγγνώμη. Κοιτάξτε, σα παρακαλώ εγκαταλείψτε την αίθουσα τη Ολομέλειας, αλλά αφήστε και του συναδέλφου να προβούν στην επεξήγηση ψήφου. Κύριε Κουντή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με το δικαίωμα θεώρησης των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων. Η πάγια θέση της αριστεράς είναι ότι είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Επομένως κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να μετακινηθεί και να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ λοιπόν συμφωνώ με την άρση των περιορισμών και του καθεστώτος θεώρησης για τους κατοίκους των Δυτικών Βαλκανίων, ψήφισα αρνητικά στη σχετική ψηφοφορία για το λόγο ότι ο τρόπος που θέτει και αναφέρεται στο κωσυφοπαίδιο αποτελεί ουσιαστικά de facto επιβεβαίωση της μονομερούς αναγνώρισής του ως ανεξάρτητου κράτους. Αυτό κατά την άποψή μου παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και την απόφαση 1244 του 99 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αποτελεί μια πρακτική με διολίσθηση σε κατεύθυνση που δεν προωθεί την ειρηνική επίλυση των διαφορών, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Κορνέλια Έρνστ για ένα λεπτό. Κυρία Κορνέλια Έρνστ είναι παρούσα? Έχω δώσει το κείμενό μου σαν γραπτή δήλωση. Καλώς σας ευχαριστώ. Μίλαν Μον. Κύριος Μίλαν Μον, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφέρομαι στην έκθεση φαγιών. Είμαι μέλο τη Ισπανική Αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματο. Θέλω να σα πω ότι εμεί υπερψηφίσαμε την έκθεση, αλλά δεν συμφωνούμε με την αιτιολογική σκέψη 2α που βάζει τροπολογία 4, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να αρχίσει διάλογο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, απαλλαγή θεώρησης από το κοσυφοπαίδιο για να ε, απελευθερωθεί το καθεστώς και να δοθούν διευκολύνσεις αντίστοιχες με τα σχέδια που υπάρχουν για άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια μοίρα το κοσφοπέδιο με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Θυμίζω ότι το Ισπανικό κράτο, οι ισπανικέ αρχέ και, καμιά, ε, και άλλες χώρες της Ένωσης δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο. Και επειδή ψηφίστηκε αμπλόκ η τροπολογία αυτή με πολλέ άλλε μαζί, εμεί δεν μπορέσαμε να την καταψηφίσουμε. Αλλά θέλουμε να σας ε, πούμε και να δηλώσουμε ότι δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μιλανμόν. Κοράτσα Μπίλτ. Για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να πω ότι η κοινή δήλωση είναι μεγάλη επιτυχία και πρέπει να το τονίσουμε. Στην κοινή δήλωση στέλνουμε ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Υποστηρίζουμε την επιτάχυνση της χορηγήσεως ελεύθερου καθεστώτος από τις θεωρήσεις στους κατοίκους των Δυτικών Βαλκανίων. Χάρη στη θέση του ΕΛΚ ξαναμπήκε σωστή τροχιά διαδικασία από σωστή κατεύθυνση και υπάρχει σωστή νομική βάση σύμφωνα με τις συνθήκες. Χάρη σε αυτό είχαμε επιτυχία. Το να έχουν πολιτική δήλωση σε ένα παράρτημα ήταν κάτι παραπλανητικό και θα έστελνε λάθος μήνυμα. Θα δημιουργούσε λάθος προσδοκίες στους λαούς της περιοχής. Εγώ ήθελα να πω ότι έζησα την πολιορκία και το βαρδισμό του Σεράγεβο για 1,5 χρόνο και είχα δεσμευτεί να επιταχυνθεί η ε, διαδικασία για να απαλλαγούν ε, ε, οι κάτοικοι της χώρας αυτής από την ανάγκη θεώρησης. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία. Ο κ. Λάιτφριντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Παλιαδέλη ε, διότι πιστεύω ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής πρέπει να εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και έγινε ε, κάτι πέρυσι το οποίο είναι τελείως αντίθετο προς αυτό το στόχο. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραπονέθηκε για ε, ένα τσίρκο που στήθηκε παρόλο που υπήρχε απαγόρευση απαγόρευση για τα άγρια ζώα δεν είναι δικιά του δουλειά υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι οι οποίοι είναι υπέρ ή κατά των τσίρκων και των αγρίων ζώων οπότε δεν νομίζω ότι αυτέ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Σας ευχαριστώ έχω τη χαρά να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία βουλευτών και άλλων επισκεπτών του Καναδικού Κοινοβουλίου και τις αντιπροσωπείες του Καναδά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πήραν θέση στο θεωρείο, το διπλωματικό θεωρείο του ημικυκλίου. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είναι στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν με τους ομολόγους τους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.